της της συνεδριάσεως. Και πριν περάσουμε στις σημερινές ψηφοφορίες, για, τις, για τα άλλα τμήματα και για τις πληρωμές, ο Γενικός εισηγητής ήθελε να επισημάνουμε μια διόρθωση στις πληρωμές των πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Ντανιέλ Διώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω όντω μια διευκρίνηση όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Χθε στην σχετική ψηφοφορία το πακέτο που ψηφίσαμε περιλάμβανε και τις πληρωμές. Το μισό δηλαδή των υποχρεώσεων συν τις πληρωμές σύμφωνα με τον κανόνα. Αλλά πρόκειται για ένα τεχνικό σφάλμα γιατί δεν τηρήσαμε τον κανόνα. Δεν ερμηνεύσαμε σωστά τον κανόνα αυτό. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτήν την τεχνική διόρθωση για τεχνικές δηλαδή τιμές που αναφέρονται στη γραμμή 04037725 8.950.000 πληρωμή, αντί για 7.905.000. Μετά στην γραμμή 3304 ε, 74 630 εκατομμύρια αντί για 507 500. Αυτές είναι οι δύο τροποποίησεις λοιπόν σχετικά με το πακέτο που εγκρίναμε χτες και ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον Γενικό Εισηγητή. Σημειώνουμε την ε, ανακοίνωση αυτή. Και θα φροντίσουμε για την σχετική διόρθωση. Καλώς, τώρα θα ψηφίσουμε τις πληρωμές. Έχουμε δύο κομμάτια. Μπορούμε νομίζω μαζί να τα ψηφίσουμε. Έτσι, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Και τώρα με κατατμήματα χωριστή ψηφοφορία, μάλλον χωριστή ψηφοφορία, έχουμε μια συμβιβαστική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Καλώς αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε έτσι τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών του τμήματος 3. Και τώρα περνάμε στα άλλα τμήματα. Άλλα τμήματα τα οποία βέβαια έχει αναλάβει ο Πολ Ρούμπικ. Αρχίζουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μπορούμε μαζί, συνολικά, μπλοκ, να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Σωστά. Αντίρρηση. Ωραία. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, στο σύνολο αυτό τροπολογιών. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τώρα. Έχουμε δύο υποομάδες που αποτέλεσαν αντικείμενο συμβιβασμού. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί. Ωραία, Τι ψηφίζουμε λοιπόν αυτές τις δύο τροπολογίες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και τώρα ερχόμαστε σε διάφορες τροπολογίες που θα πρέπει να ψηφιστούν μαζί ο σύνολο. Συμφωνείτε? Ωραία. Ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Αυτών των τροπολογιών. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Και ερχόμαστε τώρα στο establishment plant. Υπέρ. Είναι η κατά; Κατά αποχές εγκρίθηκε αυτή η τροπολογία. Ελεκτικό συνέδριο τώρα. Έχουμε μια συμβαστική πρόταση με μια υποομάδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουμε διάφορες τροπολογίες που θα πρέπει να ψηφίσουμε μαζί. Έτσι δεν υπάρχει αντίρρηση. Ωραία, τις ψηφίζουμε όλες μαζί λοιπόν, συνολικά τις τροπολογίες αυτές. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τώρα. Έχουμε εδώ πέρα συμβιβασμό σε δύο υπομπλοκ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Στη συνέχεια έχουμε διάφορες τροπολογίες που ψηφίζονται χωριστά. Η FTD 8885 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η NF 8215 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 7384 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 7385 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 7386 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 7387 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. INF 82-16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η FDD 88-86 Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FDD 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η NF 82-17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FDD 88-88 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα, συμβιβαστική τροπολογία, σου μπλοκ 1. Και έχει ζητηθεί εδώ χωριστή ψηφοφορία για το FDD 7388, λέει ο πρόεδρος. Badge 2400. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνατε. Άρα η 73-88 η FDD πίπτει, η FDD τώρα 89-83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα έχουμε τρεις τροπολογίες. ECR 8415 υπέρ. Κατά. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». EFDD 7389. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχουμε διαφορετικό κατάλογο ψηφοφοριών εδώ, αλλά νομίζω την 1420 πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε και την τροπολογία SND 7682. Πρώτα τις κάτω από το σχέδιο προπολογισμού και μετά τις άλλες. Ναι, ναι, στον κατάλογό μας λείπουν δύο τροπολογίες. Έχουμε μόνο τη δικιά μας, όλος παραδόξος. Μας λείπουν οι άλλες δύο. Λοιπόν, ε, απορρίφθηκε 84-15 λεπτο Τώρα η FDD 73-89, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. S&D τώρα, 76-82, υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Όσοι δεν έχετε ψηφίσει ακόμα ψηφίστε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε 24 ψήφοι κατά 10 υπέρ. Η FDD 7390 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 7391 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 8892 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 7392 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 8894 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η FDD 8895 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η FDD 7393 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η NF 8218 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η FDD 8896 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία τώρα. Badge 2401 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η FDD 7396 καταπίπτει έτσι. Οπότε η FDD 7397 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ECR 8416 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Η FDD 8897 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FDD 8898 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FDD 8899 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική. Σουμπλοκ 1. Μπάτζ 2402 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η FDD 7400 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. FDD 7401 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική σου μπλοκ 1, μπάτζ 2403 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η FDD 8901 καταπίπτει. Η FDD 8902 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FDD 7402 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FDD 7403 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FDD 8904 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική. σου μπλοκ 1. Μπάτζ 2404 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η FDD 7405 κατά πίπτη, η NF 8220 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 7406 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FDD 7408 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7410 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται συμβαστική σου μπλοκ 1 μπάτζι 2405 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η FDD 8905 καταπίπτει. Εξετάζουμε τώρα τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, συμβιβαστική που έχει να κάνει με δύο υπομάδες σου μπλοκ θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε μαζί. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είδα πολλά χέρια, οπότε θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίθηκε 25 υπέρ, 8 κατά. Και περνάμε τώρα στις χωριστές ψηφοφορίες επί των τροπολογιών. Η FDD 8906 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. FDD 7411 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. FDD 8907 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FD28908 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η NF8222 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FD28909 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική σου μπλοκ 1, badge 2500 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και η FTD 8910 καταπίπτει. Η FTD 8911 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 7415 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 7416 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 7417 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική σου μπλοκ 1, μπάτζ 2501 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η FTD 7418 καταπίπτει, η CR 8419 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 7419 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 7436 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 8912 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. FTD FTD 7420 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. FTD 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 7421 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 8917 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται η FDD 7423 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται συμβαστική badge ε, 2502 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η FDD 7424 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η FDD 7425 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FDD 7426 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η FTD 7427 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 7428 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η FTD 7429 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική badge 2503 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η FTD 7430 καταπίπτει. Συμβιβαστική μπάτζη 2504 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η FTD 7433 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία τώρα μπάτζη 2505 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η FTD 7434 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία μπάτζ 2506 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η FTD 7435 πίπτη Περνάμε τώρα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Χωριστές ψηφοφορίες πρώτα. Η FTD 8924 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η FTD 7500 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. EFTD 89-26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7685 και Πέτη 62-75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Νομίζω τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τι υπόλοιπε τροπολογίε EFDD απο 8128 μέχρι την 75 Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. Τώρα ερχόμαστε στο establishment plan. 56276, S&D 7686, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. επόπτης ε, προστασίας δεδομένων τώρα. Νομίζω ότι μπορούμε και εδώ να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες του EFDD εκτός από την, ε, των σοσιαλιστών, δηλαδή 7681. Οπότε ψηφίζουμε όλες τις τροπολογίες, EFDD, ENF και τα λοιπά, εκτός από την S&D 7681 που θα ψηφίσουμε Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Και τώρα ψηφίζουμε την 7681 των Σοσιαλιστών. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε δύο υποομάδες, συμβιβασμός, ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Και τώρα έχουμε τις χωριστές ψηφοφορίες. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί όλες τις τροπολογίες εκτός από την ΑΦΕΤ 5176 και την EFT 28979 και την Batch 4409. Λοιπόν, για τις υπόλοιπες που μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική τροπολογία ΦΕΤ 5176. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και η FDD 8979 και η Badger 4409 ε, καταπίπτουν. Τώρα ερχόμαστε στο Establishment Plan ε, ΑΦΕΤ 6541 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρατήρηση. Αφέτ 5176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Nous allons maintenant nous prononcer. Και τώρα συνεχίζουμε και πάμε στις πιστώσεις του τμήματος 1, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Nous avons λοιπόν, έχουμε πρώτα απ' όλα Sur, euh, les amendements Τις τροπολογίες που θα βρείτε στο παράρτημα 1 και στο πίνακα 2. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε χωριστά. Το πρώτο, το πρώτο πίνακα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Τα νέα αιτήματα τώρα των πολιτικών ομάδων. Άλντε 78-10. ΕΛΚ, SND, ΓΚΟΕ, πράσινη. Και αλτε 78 78-10 όλα αυτά θα ψηφιστούν μαζί. Πρόκειται για αύξηση της ανάληψης υποχρεώσεων ε, με ουδέτερο τον προπολογισμό, με κάποιες αντισταθμίσεις υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε χωριστές ψηφοφορίες S&D 77-91 υπέρ, κατά, αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. 18-15. Σοσιαλιστές και δημοκράτες 77-90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στα σχόλια. Γκούε 70-01 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπου 70-14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σεντή 77-90 υπέρ, κατά. Αυτό θέλει επαλήθευση, παρακαλώ, ηλεκτρονική. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται 12-20. Μπάτ 42-63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γκου 70-12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Eh bien, nous en avons Τελειώσαμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Και η ώρα είναι 9 και 37 πρώτα λεπτά. Θα ήθελα να συγχαρώ εγκαρδιότατα τους δύο εισηγητές μας, τον γενικό μας εισηγητή κύριο Ντανιέλε Βιώτη, και τον εισηγητή για τα υπόλοιπα τμήματα Παουλ Ρούμπιχ και θα σας χειροκροτήσουμε κιόλας. Mais euh, euh, Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τους γεώδεις εισηγητές και όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτές τις ψηφοφορίες και τους συνεργάτες μας που ε, προετοίμασαν τόσο άξια ε, τους καταλόγους ε, ψηφοφοριών και τους πολιτικούς συμβούλους. Peut-être que δεν ξέρω αν θέλουν να μιλήσουν οι εισηγητές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κύριε Βιώτη, θέλετε να πάρετε τώρα το λόγο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ όλος ιδιαίτερος να ευχαριστήσω ε, όλους εκείνους που συνεισέφερε στην προσπάθεια αυτή και τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους μας ε, πάρα πολύ επαγγελματικά εργάστηκαν. Καλά, αυτό το ξέρω εδώ και τέσσερα χρόνια, αλλά τώρα είχα την απόδειξη ακόμα πιο εμ, απτή. Μας βοήθησαν όσο μπορούσαμε και ε, όσο μπορούσαν ε, και εμένα και τους κοιόδης ηγητές, τους οποίους ευχαριστώ και αυτούς και ήρθε σε αίσιο πέρα στη συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας. Τώρα είμαστε στα χέρια της υψηλής πολιτικής, κύριε Πρόεδρε, ε, στο Συμβούλιο. Απέναντι στη διαδικασία της συνδιαλλαγής θα πρέπει να φανούμε όσο γίνεται πιο αποφασισμένοι. Και σε δύο εβδομάδες ελπίζω να εγκριθεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου Προπολογισμό. Απαντήσεις έχουμε και πιστικές στα ερωτήματα των πολιτών με τον προπολογισμό αυτό και απαντήσεις επίσης που αντιστοιχούν στις δικές μας αξίες και αρχές ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο, τις οποίες καλούμε θα ανακτήσουμε. Με την αντιπροσωπεία λοιπόν που θα μας υποστηρίξει και όλη την ομάδα της συνδιαλλαγής προχωρούμε σύμφωνα με τις αρχές και τις, ε, τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει στα πλαίσια μια σοβαρή διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Ελπίζω, νομίζω μάλλον ότι είναι ευνοϊκό το κλίμα και η Ιωνία. Κύριε Ρουμπίχη, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμότατα όλους. Φυσικά πρώτα απ' όλα τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω η διοίκηση εδώ έδειξε πάρα πολύ καλά ότι μπορούν να συγκεραστούν διάφορα συμφέροντα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες των πολιτικών ομάδων, γιατί έγιναν πάρα πολλές άτυπες συζητήσεις, όπως καταλαβαίνετε, και καταλήξαμε σε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δικούς μας βοηθούς και συνεργάτες, τους προσωπικούς που <laughs> μας ελέγχουν πάντα, μας κρατάνε σε ένα πλαίσιο, μας ενημερώνουν και μας βοηθούν για να ε, εργαστούμε σωστά. Αυτό ήταν τώρα το απλό κομμάτι στο ε, εσωτερικό του Κοινοβουλίου να καταλήξουμε σε μία γνωμοδότηση. Ακολουθεί το Ακανθόδες. και ε, ε, αυτό είναι η διαπραγματεύση τώρα με το Συμβούλιο. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει πάρα πολύ ήδη στις προετοιμασίες και αυτό που πρέπει να κάνει τώρα είναι να έχουμε την ίδια φωνή όλοι απέναντι στο Συμβούλιο και χαίρομαι που όλες οι πολιτικές ομάδες και ιδιαίτερα ο συνάδελφος Βιώτη έχει ε, εργαστεί πάρα πολύ εκ των προτέρων και ο Πρόεδρος. Ε, νομίζω ότι είναι κρίσιμο να είμαστε ενωμένοι απέναντι στο Συμβούλιο για να επιτύχουμε. Το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να δείχνει το δρόμο, να ανοίγει το δρόμο και χαίρομαι εγώ και για την τριμερή διαπραγμάτευση και τη συνδιαλλαγή. Ξέρω ότι εύκολο δεν θα είναι, αλλά είμαστε πολύ αποτελεσματικοί σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Merci. Merci. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά για τα λοιπά τμήματα. Και πάλι ισχύει σαν για άλλη μια φορά στο κοινοβούλιο. Euh, euh, euh, Τα κράτη-μέλη, όταν είναι ενωμένα, ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν ισχυρά την ε, παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις της. Τώρα, θα ήθελα να δώσω λόγο στον κύριο Γιώχαν Ιουρέλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρώτα μπορώ να τον συγχαρώ, διότι ορίστηκε διευθυντής. Άξιος επάξια αναγνώριση. Ο μας <laughs> Και μια που έχετε την τιμητική σας, μήπως έχετε και κανένα σχόλιο για την ψηφοφορία και το αποτέλεσμά της εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια ε, και τα εκτιμώ πάρα πολύ. Σύντομα. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Βιώτη και τον κύριο Ριμπίχ, τους συζητητέ. Ήταν ε, πολύ περίπλοκη δέσμη αυτή. Εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είμαστε εκτός γηπέδου και σας περιμένουμε και εσείς συνήθω δυσκολεύεστε, αυτή τη φορά έγιναν όλα πάρα πολύ απρόσκοπτα και αυτό είναι εξαιρετικό ιονός για το μέλλον από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά τα ειλικρινή μα συγχαρητήρια για την επιτυχία αυτή. Γενικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που ενέκρινε πολλές τροπολογίες που επαναφέρουν τα ποσά ε, ε, ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμών που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο και πολύ καλή αφετηρία για τη συνδελαγή. Πάρα πολύ σύντομα κάποια ειδικά σχόλια. Προφανώς θα επανέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Σε ό,τι αφορά το τίτλο 1α, είναι σαφές ότι η εστίαση των διαπραγματεύσεων θα αφορά πάρα πολύ το Erasmus Plus, Erasmus Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο Ε, ψήφισε αυξήσεις ε, στην κατηγορία αυτή, στον τίτλο αυτό και τα δύο τρίτα των αυξήσεων αφορούν το Erasmus Plus και το Erasmus Youth, την νεολαία. Βέβαια, το Συμβούλιο από την πλευρά του ε, δεν προχώρησε σε μειώσεις στο Erasmus και περικοπές και είναι από τα λίγα προγράμματα το δεν το έκανε αυτό. Ε, είναι καλό σημάδι λοιπόν που θεωρούν προτεραιότητα και τα δύο σκέλη της Δημοσιονομικής Αρχής στο πρόγραμμα Εράσμος. Ε, στο τίτλο Β θα κυριαρχήσει ένα θέμα, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνουμε την ψηφοφορία σας για σημαντική αύξηση της πρικοδότησης αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι θα είναι δύσκολη η συζήτηση με το Συμβούλιο. Ιδιαίτερα αν η προτινόμενη αύξηση υπερβαίνει τα ποσά που συμφωνήθηκαν στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτές του δημοσιονομικού πλαισίου πριν από δύο χρόνια. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως διαμεσολαβητής για να σας διευκολύνουμε να συμφωνήσετε. Θα πρέπει να επαναλάβουμε την ανησυχία μας ότι η αύξηση ε, των κονδυλίων για, για την απασχόληση των νέων δημιουργούν και κάποιες νομικές υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη ε, για μια αντίστοιχη αύξηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις γραμμές του προϋπολογισμού και υπάρχει κίνδυνος να έχουμε καθυστερήσεις ε, στην εκτέλεση των πόρων του Ταμείου αυτού, του Κοινωνικού Ταμείου. Τα ξέρετε αυτά. Σημειώνουμε την πολιτική προτεραιότητα που συνιστά αυτό το θέμα για το Κοινοβούλιο και σίγουρα θα κυριαρχήσει και στη συνδιαλλαγή σε ό,τι αφορά ε, τον τίτλο 2 και τη γεωργία. Μέσα Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την ε, παραδοσιακή τροποποιητική επιστολή στον προπολογισμό και θα περιλαμβάνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για ε, τη Γεωργία και θα έχει την ευκαιρία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει μια ενημερωμένη εκτίμηση όλων των αναγκών και βέβαια και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις όπως είναι ε, η έξαρση και τα κρούσματα της αφρικανικής πανόλης του χείρου που έχουμε σε διάφορα κράτη-μέλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης που επαναφέρατε τα ποσά και σβήσατε κάποια αποθεματικά που ως μη όφιλε το Συμβούλιο έχει γράψει, ας πούμε για το Δουβλίνο, Ξέρουμε ότι είναι πολύ κρίσιμε οι διαπραγματεύσει, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να δεσμεύουμε κονδύλια και να τα βάζουμε και σε ένα αποθεματικό. Ε, σας ευχαριστώ. Ε, στον τίτλο 3 οι ανάγκε επίση μεταβάλλονται συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το παρακολουθεί και θα δούμε μέχρι τη συνδιαλλαγή αν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να ε, προτείνουμε ε, αυξήσεις τροποποιητική μας επιστολή μέσα Οκτωβρίου μπορεί να προτείνουμε κάποια νέα στοιχεία σχετικά. Ε, Στον τίτλο 4 ε, και πάλι το βασικό θέμα συζήτηση, όχι το μοναδικό, θα είναι ε, το πρωταξιακό μέσο και σε σχέση με την Τουρκία και το πώ χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό οι για του πρόσφυγε στην Τουρκία. Δεν θέλω να πω στην ουσία αυτού του τόσο ευαίσθητου και λεπτού θέματο σήμερα, αλλά επειδή έχω ζήσει αυτές τις συζητήσεις στο Συμβούλιο μήνες ολόκληρους, δεν θα σας αποκαλύψω κανένα μυστικό λέγοντας ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ το Συμβούλιο να κινηθεί στο θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές δαπάνες, θέλω να σας ευχαριστήσω, ιδιαίτερα τον κύριο Βιώτη που προτείνει και την Επιτροπή που δέχτηκε να επανέλθει ε, το επίπεδο ε, του σχεδίου προπολογισμού που προτείναμε για την ανάληψη υποχρεώσεων. Οι περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο θα ε, έπληταν πάρα πολύ σφοδρά την ε, λειτουργία της διοίκησης μας. Όπως κάθε χρόνο θα σας δώσουμε λεπτομερή σχόλια στην επιστολή εκτελεσιμότητας και προς εσάς και προς το Συμβούλιο επιστολή που θα σας στείλουμε πολύ γρήγορα ε, μετά την έγκριση της επίσημης θέσης του ε, Κοινοβουλίου τέλη Οκτωβρίου γύρω στις 26 του μηνός. Ε, ολοκληρώνω, Πρόεδρε και αγαπητοί εισηγητά. Με συγχαρητήρια και προς τους δύο εισηγητές φυσικά και πάλι για την τόσο επιτυχή ψηφοφορία. Αναμένονται ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις στη συνδιαλλαγή που θα μπουν και στην ουσία ε, πολλών σημαντικών θεμάτων και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πάντα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε μια συμφωνία και να κάνουμε προτάσεις όταν θεωρούμε ότι είναι χρήσιμες ε, ως ε, έντιμος και ειλικρινής διαμεσολαβητής. Ευχαριστώ πολύ. Merci, le directeur. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά, τόσο μας είπατε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση της Κομισιόν στην προσπάθεια εξέβρεση μια συμβαστική λύση με Επιτροπή και Συμβούλιο. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Όσον αφορά το amending letter, 26 Οκτωβρίου λοιπόν, ή 15 ποια είναι, α, με διορθώνουν, και η επιστολή εκτελεσιμότητας. Έχετε κάποιες ημερομηνίε ως προς αυτό. Λοιπόν, για την ε, την ε, συνδυαλλαγή. Θυμάστε πέρσι είχαμε φτάσει και στην διαμαρτυρία ως κοινοβούλιο. Θα δούμε τι θα γίνει με τη συνδυαλλαγή, την τελευταία συνδυαλλαγή πριν το τέλος αυτής της εντολής. Αυτής της θητείας. Ευχαριστώ κύριε Ρέλ για τις διευκρινήσεις. Ε, να θυμίσω τα επόμενα βήματα ψηφορία 8 και 9 Οκτωβρίου, τριμερής διάλογο 18 Οκτωβρίου, συζήτηση στην Ολομέλεια της θέση 23 και 24 Οκτωβρίου, έναρξη της συνδιαλλαγής πρώτη συνδρίαση 7 Νοεμβρίου, δεύτερη, ελπίζουμε, θα είναι και τελική, 16 Νοεμβρίου και η τελική. Τελική. Ελπίζω να τελειώσει λογική ώρα. Πολύ ωραία. Και Γιώργης αν ήταν εδώ θα του είχα δώσει το λόγο αλλά κολλείεται μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω είχε προετοιμάσει έκθεση σχετικά με αυτό το οποίο ονομάζουμε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων μεταξύ των προτάσεων του κ. Γκέρενς διαβάζουμε τη διαπίστωση περί άκρη του πολλαπλασιασμού των ταμείων, κάτι το οποίο καθιστά δυσανάγνωστο τον προϋπολογισμό, κάτι το οποίο αντιβαίνει στο ενιαίο του προϋπολογισμού και το οποίο αποδεικνύει αυτό το οποίο είχε υπογραμμίσει η έκθεση Μόντι περί ενός γαλαξία ταμείων και ενός δημοσιονομικού γαλαξία που καθιστά δύνατη την ανάγνωση, την ευλογή ανάγνωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Ένωση. Προτείνει ο κύριος Γκέρενς να μειώσουμε αυτόν τον αστερισμό προπολογισμών και ταμείων στο πλαίσιο και του πίδελταπή και μέσω μιας τακτικής νομοθετικής διαδικασίας. Επιμένει μάλιστα όσον αφορά την ανάγκη ψηφορίας με τη βάση της ειδικής πληψίας και όχι της ομοφωνίας στο Συμβουλίο. Και τούτο για τον εξορθολογισμό της υλοποίησης του προϋπολογισμού για να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αποφάσεων που αφορούν την ουσία της Ένωσης και να αποφύγουμε και τις πατάλες. Και υπογραμμίζει επίση. τη λειτουργία της Γερμανικής Βουλής πριν την επανένωση, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Λαμβάνουμε λοιπόν επίσης και του, τις ψήφους της περιφέρειας. Δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη επιπλέον οι ψήφοι των χωρών που εμπλέκονται στο α στο β πρόγραμμα. Έστω και με συμβουλευτικό τρόπο. Για τα επενδυτικά στρατηγικά ταμεία πρέπει επίση να ληφθούν υπόψη οι συντελεστέ, οι δείκτε αποτελεσματικότητα, οι εθνικέ συμμετοχέ, έτσι ώστε τα κριτήρια κατανομής των σχετικών πόρων να βασίζονται στην τήρηση, να εξαρτώνται από την τήρηση από τα κρατημέλη των κανόνων τη ελληνική, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη δίκαιης κατανομής των αρμοδιοτήτων και ευθυνών. η ουσία τη έκθεση. Λοιπόν, είναι αυτές οι προτάσει, αυτέ οι συστάσει είναι οι συστάσει και οι προτάσει του συναδέλφου Γκέρεν. Ο λόγος στο Κιώδης στον κύριο Ντοσάντο πρώτα, ο οποίο δεν είναι εδώ. Θέλει κανεί τον λόγο για να σχολιάσει τις προτάσεις Γκέρεν. Κανεί. Πολύ ωραία. Τον συγχαίρω. Διευκρινίζω ότι οι τροπολογίε επί του σχεδίου έκθεσης πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στι 11 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 5 Νοεμβρίου και η ΑΦΚΟ. Ψηφίζουμε 21 Νοεμβρίου. Θα δώσω τώρα τον λόγο στους συναδέλφους που συνέγραψαν γνωμοδότηση για τα διάφορα προγράμματα του επομένου ΠΔΠ. Ο λόγος πρώτα απ' όλα στην κυρία Γιάτεν Μάκη, πρόγραμμα για το περιβάλλον, για τη δράση, για το κλίμα. Ανελή, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, συνάδελφοι, καλημέρα. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι για την πρόταση της Κομισιόν, γι' αυτό και δεν χρειάστηκε να υποβάλω πολλές τροπολογίες. Επίσης, μου άρεσε και η υπόφαση των συντονιστών να μειώσουμε το πεδίο επανεξέταση των δημοσιονομικών ε, θεμάτων. Πρόκειται για το μόνο πρόγραμμα το οποίο αφορά το κλίμα, το οποίο χρηματοδοτεί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιβάλλον και το κλίμα. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στους δύο αυτούς τομείς είναι τεράστιες κλίμακα, είναι παγκόσμια προβλήματα και συναφώς απαιτείται συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν τούτου δικαιολογείται πιστεύω να αυξήσουμε τον σχετικό προϋπολογισμό του προγράμματος του LIFE. Με βάση αυτά τα οποία έχει δηλώσει το Κοινοβούλιο, προτείνω το ανώτερο όριο να διπλασιαστεί σε σχέση με τα εφιστάμενα επίπεδα. Εσωτερικά, όσον αφορά την κατανομή, δηλαδή των πόρων, το πρόγραμμα διαιρείται σε δύο κλάδους δραστηριοτήτων πρώτος αφορά το περιβάλλον. Το δεύτερο αφορά τις δράσεις για το κλίμα. Και μετά όλα αυτά διορούνται σε υποπρογράμματα. Πρέπει να ενισχύσουμε, να αυξήσουμε τις ε, πιστώσεις και για τα δύο προγράμματα, αλλά η χρηματοδότηση να δώσει έμφαση μάλλον στο περιβάλλον. Με τις τροπολογίες προτείνω 70% να πάνε στο περιβάλλον και 30% στις δράσεις για το κλίμα. Στην πρόταση της Κομισιόν τα αντίστοιχα ποσοστά είναι ελαφρώς διαφορετικά, είναι 64 περίπου, 64 και 36%. Όσον αφορά τα υποπρογράμματα, κάθε κλάδου, κάθε. Προτείνω να δεχθούμε την κατανομή που προτείνει η Κομισιόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να αποφύγουμε παρανοήσεις, να καταστήσω σαφές εξ αρχής ότι η πρότασή μου δεν αποσκοπεί στην ακύρωση της ανάγκης χρηματοδότησης των δράσεων για το κλίμα. Το αντίθετο, προτείνω να παραμείνει η ίδια, η ε, ίδια η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα στο επόμενο πηδελταπή 30%. Όμως, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι εντός του LIFE τροποποιούμε ελαφρώς την ε, κατανομή για να ενισχύσουμε άλλους στόχους για το περιβάλλον, δεδομένου ότι οι δράσεις για το περιβάλλον θα χρηματοδοτηθούν και από άλλα προγράμματα στο επόμενο ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Κάτι το οποίο δηλαδή δεν συμβαίνει από την άλλη μεριά για τα προγράμματα για το περιβάλλον καθαρά. Γι' αυτό και το περιβάλλον χρειάζεται ενίσχυση. Πρώτο βλέπω στα σχόλια των σκιωδών εισηγητών και των άλλων συναδέλφων και θα χαρώ πολύ να συνεργαστούμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε εισηγητρία. Εισηγητές. Κύριε Λαβιά. κύριε Καπούτο. Χαίρομαι για την πρόταση της Κομισιόν, εκφράζω την ικανοποίησή μου. Σύρκα με το live και το επόμενο πί. Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδεικνύει την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστιμένη αξία της. Είμαι υπέρ τη αύξηση των πόρων για το Life 60%, αν και αυτό δεν είναι αρκετό, κατά τη γνώμη μου. Χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια. Είναι το μόνο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ακριβώς αφορά του στόχου για το περιβάλλον και το κλίμα. Χρειάζεται επίση να διευρύνουμε το αντικείμενο και τους στόχους του προγράμματος. Ε, πρόκειται για στόχους τους οποίους το σημερινό ΠΔΠ τους έχει στο Horizon. Διάβασα και τις τροπολογίες της κυρίας την Μάκη, τη συγχαίρω. Η θέση της είναι λίγο πολύ και η δική μου θέση και η θέση της NV. Το 70-30, 70 για το περιβάλλον και 30 για τις δράσεις για το κλίμα αφορά τα 7,3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τα σχετικά προγράμματα. Θα αξιοποιήσουμε έτσι τις διαθέσιμες πιστώσεις με τον κατάλληλο τρόπο σε συνεργασία και με το Περιφερειακό Ταμείο. Χρειάζεται όμω ενημέρωση, χρειάζεται τεχνική βοήθεια για να βοηθήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τους πόρους. Έχει σημασία λοιπόν επίση η δικτύωση με τα εθνικά σημεία επαφής, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η διεθνή συνεργασία. Τέλος, συμφωνώ με την ανάγκη να κινητοποιήσουμε κεντρικούς και για το περιβάλλον. Χρειάζεται όμως ε, να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τις ε, μικτές χρηματοδοτήσεις και αυτό πρέπει να το καταδείξουμε μέσω πιλωτικών προγραμμάτων όπως έγινε και στην περίοδο 2014-2020 στα πλαίσια του Live. Πρόεδρος, άλλος που θέλει το λόγο. Κυρία Γιάτεν Μάκη, Έχετε την υποστήριξη της Επιτροπής μας, προπολογισμών, τροπολογίες, 12 ώρα το αργότερο, 1η Οκτωβρίου. Η ψηφορία σε εμά θα γίνει 5 Νοεμβρίου. Κατόπιν τούτου, είναι το λόγο στον πρόεδρό σας, ο οποίος είναι εισηγητής για το Έρασμό Συν. Να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι το είναι ένα εμβληματικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των νέων Γιορτάσαμε τα 30 χρόνια, το 2017, 30 χρόνια του Εράσμος. Ένα σωρό νέοι, 6 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια νέοι είχαν χάρη στο αρισμό στη δυνατότητα να μεταβούν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανακαλύψουν ακριβώς την πολυφωνία της Ένωσής μας. Έμαθαν ξένες γλώσσες, τελειοποίησαν τις γνώσεις τους σε ξένες γλώσσες εκτός από την μητρική τους γλώσσα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Το πρόγραμμα που μας προτείνει η Κομισιόν είναι ικανοποιητικό. Το ερώτημα είναι όμως, είναι επαρκείς οι πιστώσεις, τις βρίσκουμε επαρκείς. Όπως γνωρίζετε, εδώ υπάρχει και απογοήτευση διότι μόνο μία στις δύο επιλέξιμες αιτήσει εν τέλει ικανοποιείται. Ελήψη πιστώσεων. Θα θέλαμε επίσης το έρασμος να μην περιορίζεται μόνο στους φοιτητέ. Θέλουμε το έρεσμος να καλύψει και μαθητευόμενους επαγγελματική κατάρτιση. Διότι αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι για την ενεργεία των νέων στην Ευρώπη, που πλήττει κατά κύριο λόγο συγκεκριμένες χώρες, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι χώρες οι οποίες έχουν παράδοση στην επαγγελματική κατάρτιση δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα ενεργείας. Λοιπόν, θα ήταν καλό να διευρυνθεί η μαθητεία, ο θεσμός, και ποιο είναι το καλύτερο εργαλείο, αν όχι το έρασμος. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε σε όλες τις χώρες και τις κυβερνήσεις να κάνουν στόχο την επαγγελματική κατάρτιση βάσει και συμβάσεων εργασίας, τα μεικτά συστήματα. Γιατί πολλές φορές η εθνική νομοθεσία δεν διευκολύνει αυτή την μεικτή ε, μαθητεία Πολλέ φορέ μάλιστα περιορίζει και τι δυνατότητε μετακίνηση Περιορίζει την κινητικότητα. Πρέπει λοιπόν ε, να, είμαστε στην υπηρεσία των νέων, να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά του, να ενισχύσουμε το πρόγραμμα, προσθέτοντα λοιπόν δυνατότητε και για του μαθητευόμενου και όσου ε, συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματική κατάρτιση. Στην έκθεση πρωτοβουλία τη κυρία Τωμά και του κυρίου Όλμπριχτ τον Μάρτιο προτάθηκε να πολλαπλασιαστούν επί τρία τα κονδύλια για το αρισμό. Και το πιστεύω αυτό. Προτείνω λοιπόν και υποβάλλω τροπολογίε, σύμφωνα με τι οποίε θα αυξηθούν όλες οι πιστώσει του προγράμματο. Και επιμένω επί του εξή πράγματο. Το ετήσιο πρόγραμμα, όπω θα προτείνει η Κομισιόν σημαίνει ότι το 2021 οι θα είναι μικρότερες από αυτέ του 20, του 2020. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν με να επαναθεωρήσει τους πόρους στο πλαίσιο του ΠΔΠ και να φροντίσει το 2021 σε καμία περίπτωση να μην πέσουμε κάτω από τα κονδύλια του 2020 για το αερασμός. Γιατί θα προκληθεί καταστροφή η οποία θα είναι και ακατανόητη για τους ενδιαφερομένους. Όπως είπα, συμπεριλαμβάνουμε επίσης στους δικαιούχους όσους συμμετέχουν σε επαγγελματική κατάρτιση και σε πρόγραμματα μαθητείας Αύξηση λοιπόν σε σχέση με την περίοδο 14-20. Όσον αφορά τον έλεγχο, να τονίσω το εξή. Οι έλεγχοι μειώθηκαν. και αποτελούν σήμερα ένα δυσανάλογο εμπόδιο. Θα ήθελα λοιπόν οι έλεγχοι να επαναπροσδιοριστούν και να περάσουν στα χέρια της κάθε σύμφωνα με τους εκεί δημοσιονομικού κανόνες. Διότι χθε συναντήθηκα με την Γαλλία υπεύθυνη για το έρασμό και μου είπε ότι έγιναν στη χώρα τη πέντε έλεγχοι μέσα σε ένα χρόνο για το έρασμό. Πέντε έλεγχοι. Μιλάμε λοιπόν για απλούστευση. Θα ήθελα τα προγράμματα να συλλειτουργήσουν και όχι το καθένα ανεξάρτητα. Και το λεφτό γιατί διαπιστώσαμε ότι η Γενική Διεύθυνση απασχόληση, είχε άλλους κανόνες από τη Διεύθυνση για τον Πολιτισμό κλπ. Άλλοι κανόνες και στο πεδίο. Μια κατάσταση εξαιρετικά πολύπλοκη, ακατανόητη και του χρόνου Ξέρετε, έχουμε ευρωεκλογέ. Οι πολίτε μα έχουν ακούσει τόσο πολλά για την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, πράγμα το οποίο είναι ακόμα ακατανόητο και βεβαίω απαράδεκτο εκφράζω την, ε, τον ευσεβή ενδεχομένω πόθο οι διοικητικέ διαδικασίες να απλουστευθούν σημαντικά. Ο λόγος στον κύριο Νοβακόφ και ο δισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον ενθουσιασμό που δείχνετε για αυτά τα θέματα. Πραγματικά είναι έμπνευση για μας. Θέλω να αναφερθώ στον αέρα, στο πρόγραμμα Erasmus, σαν ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα γνωστό ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βελτιώνει τη ζωή των νέων όσο κανένα άλλο πρόγραμμα δεν το είχε κάνει πριν. Υπάρχουν πολλές στατιστικές αυτά τα 30 χρόνια ιστορίας του Έρασμους. Το πιο βασικό είναι όμως να ξέρουμε ότι το 80% όσων συμμετείχαν στο Έρασμος έχουν ηγετικέ θέσεις στο χώρο εργασίας τους. Το 1 τρίτο όσων συμμετείχαν στο Εράσμους επίσης δημιούργησαν τη δικιά τους επιχείρηση. Άρα δεν καταπολεμούμε με το Εράσμους μόνο την ανεργία, δημιουργούμε και επιπλέον θέσεις απασχόληση από τους ανθρώπους αυτούς που συμμετείχαν στο Εράσμους. Το μόνο το οποίο δυσκολεύει το πρόγραμμα είναι ο προπολογισμός, η προκοδότησή του. Και αν βρεθεί χρηματοδότηση για τόσο πολλές και διαφορετικές πρωτοβουλίες, εγώ δεν θέλω τώρα βέβαια να βάλω σε αντιπαράθεση τη μία πρωτοβουλία με την άλλη, αλλά πηγαίνετε να μιλήσετε με ένα φοιτητή και να του πείτε ότι αυτός δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Εράσμους γιατί πρέπει να έχουμε έναν παραπάνω συνοριοφύλακα στα σύνορα. Δεν πρέπει έτσι να πηγαίνει. Το Εράσμους είναι ότι καλύτερο έχει συμβεί στους νέους τα τελευταία χρόνια και για μένα πρέπει να κάνουμε τα Πρώτον, go global στο μέλλον. Δηλαδή, μην μένουμε μέσα στη φούσκα μας ε, που ξέρουμε ότι προσφέρουμε καλή εκπαίδευση κτλ. Αλλά αν δείτε γενικότερα την αγορά εκπαίδευσης και σπουδών, πολλοί προτιμούν να πάνε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Άρα ας κοιτάξουμε και γύρω μας λιγάκι, ας δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους νέους Ευρωπαίους να πάνε και εκτός Ευρώπης. Υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα πριν από δύο χρόνια που είναι για τους νέους επιχειρηματίες και ήδη έχουμε 200 που έχουν συμμετάσχει και που αποφάσισαν να επωφεληθούν από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και να πάνε στη Silicon Valley, στη Σιγκαπούρη και στο Ισραήλ. Γιατί αυτές οι χώρες έχουν προχωρήσει περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιους τομείς. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, ακόμα υπάρχουν ε, γραφειοκρατικά εμπόδια και στηρίζω τον πρόεδρο. Εγώ αναρωτιέμαι πάντα πώς είναι δυνατόν αν αποφασίσεις να πας στο εξωτερικό και να χρησιμοποιήσεις την υποτροφή Εράσμους να περάσει εξετάσεις και ό,τι χρειάζεται μετά δεν αναγνωρίζετε το διπλώμά σου πίσω στη χώρα σου ή κάποιες από τις εξετάσεις δεν αναγνωρίζονται και πρέπει να τις ξαναπεράσεις. Αυτά τα μικρά πραγματάκια είναι όμως που αμαυρώνουν κάπως την λαμπρή εικόνα του προγράμματος Έρασμος. Νομίζω ότι αυτά μπορούμε να τα διορθώσουμε. Ζητάει 40 δισεκατομμύρια ο εισηγητής. Είναι κάτι το οποίο στηρίζω. Πρόκειται για επένδυση που κάνουμε και από την οποία θα έχουμε απόσβεση πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Νοβακόφ για τη στήριξή σας. Ο κύριος Σόρβας τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ και η ομάδα μου ε, σας ευχαριστεί για την έκθεση αυτή. Για την φιλοδοξία που αντικατοπτρίζει αυτή η έκθεση όσον αφορά το πρόγραμμα Έρασμος. Όντως, πρέπει τα ωραία λόγια που λέγονται για το Έρασμος να αντικατοπτρίζονται όμως και στον προπολογισμό, δηλαδή στις δημοσιονομικές προτάσεις για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχει κάνει σχετικό ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα λέμε αυτά από το Μάρτιο. Πρόεδρε, ξέρω ότι στηρίζετε τους νέους και όχι μόνο στα πανεπιστήμια και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι για αυτή την πτυχή του προγράμματος που πάει δηλαδή πιο πέρα. Και είναι απόλυτα λογικό σε μια εποχή διεθνών αλυσίδων προμήθειας νέων τεχνολογιών, η μαθητεία, η άσκηση των νέων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Οι εξελίξεις στο κατασκευαστικό τομέα στο μέλλον θα είναι διασυνοριακές, διεθνείς. Άρα είναι απόλυτα λογικό και ουσιαστικό να υπάρχει διασυνοριακή και διεθνή συνεργασία όπου να συμμετέχουν όλοι όσοι αποφασίζουν για το μέλλον. Ελπίζω και εγώ ότι το αερασμό θα μπορέσει να αντικατοπτρίσει και να στηρίξει αυτή την κατάσταση στο μέλλον. Υπάρχει το άρθρο 16 που μιλάει για τη συμμετοχή τρίτων χωρών. Η συνεισφορά και η συμμετοχή αυτών όμως θα πρέπει να είναι ανάλογη και στον προπολογισμό και να υπάρχει διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το από πού έρχονται τα χρήματα. Πλήρης διαφάνεια για όλα τα προγράμματα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσω και εγώ να εμπλουτίσω το κείμενο και με την στήριξη των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Να ληφθεί και αυτό υπόψη για το μέλλον. Επίσης χαίρομαι για αυτό που λέτε για το επίπεδο γραφειοκρατίας που πρέπει να μειωθεί στο πρόγραμμα. Και στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια έχει εκφραστεί αυτή η ανησυχία, οπότε χαίρομαι που το έχετε συμπεριλάβει. Πρόεδρος, σε ευχαριστώ. Άλλος κανείς που θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ωραία, θα καταλήξω στα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο συναδέρφους για τα σχόλιά τους και που μας στηρίζουν. Θα επανέλθω σε κάτι που ανέφερε ο κύριος Νοβακόφ, δηλαδή την αναγνώριση των κεκτημένων της κινητικότητας. Για τους φοιτητέ πάνε αρκετά καλά τα πράγματα γιατί τα πανεπιστήμια είναι οι κατάλληλες αρχές ε, για τα διπλώματα. Για την επαγγελματική όμως κατάρτιση, την ε, μαθητεία, είναι οι εθνικές αρχές. Είναι τα Υπουργεία Εθνικής Εκπαίδευσης ή τους πάντων άλλα τα οποία είναι οι αρμόδιες αρχές. Οπότε, αν ένας νέος για έξι μήνες πάει σε μια άλλη χώρα, ό,τι θα έχει μάθει εκεί, η εμπειρία που θα έχει αποκτήσει, είναι πράγματα τα οποία θα αναγνωριστούν όταν θα πάρει το δίπλωμά του στην χώρα προέλευσής του. Οπότε, αν συμφωνείτε, θα υποβάλω μία επιπλέον τροπολογία για να επιστήσω ακριβώς την προσοχή του Συμβουλίου στην αναγκαιότητα να προβεί στην αναγνώριση όλων αυτών των αποκτηθέντων προσόντων κατά τη διάρκεια της όποιας μαθητείας. Κατά τα άλλα είναι σίγουρο ότι πρόκειται για επένδυση. Το πρόγραμμα Εράσμους είναι επένδυση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Οι πρέπει να υποβληθούν πριν στις 4 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε 5 Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σόλε για τα δικαιώματα και τις αξίες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, Αυτό το πρόγραμμα για τις τα δικαιώματα και τις αξίες είναι και πάρα πολύ επίκαιρο και ε, κάτι που χρειαζόμαστε πηγόντως. Σήμερα βλέπουμε κάποια κινήματα, ακόμα και κυβερνήσεις να στρέφονται κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών, των οποίων ε, έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακόμα και την ίδια την ιδέα αμφισβητούν των ανοιχτών κοινωνιών ε, και χωρίς αποκλεισμούς, χρησιμοποιώντας λαϊκισμό, αυταρχικές ε, συμπεριφορές, ακόμα και πολιτικές. Of some, uh, οι λεγόμενες πλέον ανελεύθερες δημοκρατίες είναι αυτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά προσκρούν σαφέστατα ε, με τις ε, ε, βασικές αρχές και θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πρόγραμμα γιατί προέκυψε, γιατί υπάρχουν διάφορες ανισότητες και διάφορες διακρίσεις ε, ε, σε ευρύτατη κλίμακα και παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς υπάρχει ανάγκη να σφύρει, λατηθεί μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα που να βασίζεται σε κοινέ αξίες. Κατά την άποψή μας λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θεωρούμε ότι έχει σημασία και το επενθυμίζουμε οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ να ενσωματωθούν σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε όρους δημοσιονομικούς και πόρους που αφιερώνονται σε αυτό το πρόγραμμα προτείνουμε μια μικρή αύξηση των πόρων που συνάδει και με τον στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 1,3% του ΑΕΠ για τις επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι τρεις λοιπόν εδώ οι κλάδοι αυτού, του, αυτού του ανανεωμένου προγράμματος, τρεις πυλώνες, ε, ισότητα και δικαιώματα, συμμετοχή των πολιτών και το τρίτο είναι το πρόγραμμα Δάφνη. Με άλλα λόγια, σε αντίθεση με την αρχική πρόταση, εμείς προτείνουμε μια σαφή πρικοδότηση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Για λόγους σαφήνειας τα λέω αυτά, αλλά και για λόγους ε, συμπερίληψης της διάστασης του φύλου που λείπει πάρα πολύ από τις προτάσεις για το νέο PDP. Θα πρέπει ε, η πολιτική αυτή να συνοδεύεται και από διαφάνεια αλλά και από συγκεκριμένα ποσά στις αντίστοιχες γραμμές ε, κονδύλια του προϋπολογισμού για να ε, καταπολεμηθεί ε, η έμφυλη βία και οι διακρίσεις με βάση το φύλλο. Γι' αυτό ζητούμε να υπάρξει ρητή αναφορά και πρικοδότηση του κλάδου Δάφνη, του προγράμματος αυτού που καταπολεμά τη βία κατά των γυναικών. Επίσης, θέλουμε ε, να τονίσουμε ότι χρειάζεται να βελτιωθεί και η ποιότητα των δαπανών. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για να φτάσουμε στους στόχους αυτού του προγράμματος με ε, την καλύτερη δυνατή ε, αξιοποίηση των οικονομικών πόρων. Θα κάνω και άλλες προτάσεις ως ηγητής. Τροπολογίες, ναι, θα καταθέσω δηλαδή. Αλλά βασικά αυτά ε, είναι τα κυριότερα σημεία και οι ουσιαστικότερες προτάσεις που έχουμε συμπεριλάβει στη γνωμοδότησή μας και περιμένω να ακούσω και τους κοιόδης συζητητές και τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Ο κύριος Κωνσάλης Πόνς απουσιάζει, ο κύριος Φερνάντης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Eh, Ο συνάδελφος Κονσάλεθ Πόνς είναι δικαιολογημένος απόν και σας ζητάει συγγνώμη. Ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή. Ε, θεωρεί ότι τέτοιου είδους προγράμματα που έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά τους στην πράξη πρέπει να συνεχίζονται με την απαραίτητη χρηματοδότηση. έχουν αυτά τα προγράμματα. Αυτό δεν σημαίνει για πλούστευση. Ε, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα το υποστηρίζαμε. Αλλά θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση πλέον θα πρέπει να συνάδει απολύτως με τις προτεραιότητες όλων των θεσμικών οργάνων και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση στο Κοινοβούλιο, 1,3% του ΑΕΠ. Και αυτό το ποσοστό δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο, δεν είναι τυχαία τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά είναι αυτό που χρειάζεται για να φτάσουμε στους στόχους μας θα συνεργαστεί ο κύριος Κονσάλεθ Πόνς με τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις για να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση όπου να εκφράζονται οι ανησυχίες μας ως προς το δημοσιονομικό σκέλος αυτής της πρωτοβουλίας. Να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντς. Η κυρία Γκουαρδία Σάβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε γενικά συμφωνούμε αρκετά με την τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Απλώς εγώ έχω μια μικρή αμφιβολία ε, γιατί χωρίζονται σε δύο κονδύλια η ισότητα ε, από τη μια και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Δηλαδή είναι νεό το ποσό, γιατί το σπάτε στα δύο. Για λόγους θεματικούς, για να δούμε ότι υπάρχουν δύο κλάδοι το καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να καταδείξετε το περιεχόμενο, αλλά μια φορά όταν περιορίζουμε τόσο πολύ το πλαίσιο, ε, περιορίζουμε και την ευελιξία. Γενικά δεν διαφωνώ, απλώς θέλω να το ξανασκεφτούμε. Ε, κατά τα άλλα συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει το λόγο. Κυρία Γιάννη Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον ενισχύετε. Εξαιρετικές ιδέες σας. Τονίζω και εγώ ότι χρειαζόμαστε προπολογισμό για να ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους για τα δικαιώματα και τις αξίες. Όλο μάλλον σήμερα. Δεδομένου ότι είμαστε μάρτυρες εξελίξεων σε ορισμένα κράτη-μέλη που θίγουν το κράτος δικαίου. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα για το πρόβλημα. Εν ε, ε, δεν έχουμε τροπολογίες, ε, θα δούμε αν ε, σκεφτούμε κάτι για να βελτιώσουμε ακόμη το κείμενο. Είναι καλό πάντω το κείμενο έτσι όπω είναι. Ευχαριστώ κύριε Γιατρινάκη. Άλλο για την έκθεση του κύριου Σολέ. Όχι. Λοιπόν, τροπολογίες, κατάθεση τροπολογιών ω τι 3 η ώρα 3 Οκτωβρίου. Ψηφορία σε εμά 5 Νοεμβρίου. Κύριο Αλή για το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της απάτης. Πρώτα ευχαριστώ από τη συνάδελφη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την δημιουργία του προγράμματο για την καταπολέμηση τη με δύο βασικού στόχου. Πρώτον, προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση και δεύτερον, υποστήριξη στο πλαίσιο τη αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των ελληνικών υπηρεσιών των χωρών και τη Κομισιόν. Είναι δεδομένο ότι οι παρατυπίες και απάτη επηρεάζονται οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, αλλά φύγονται και τα κρατη Έτσι, το νέο πρόγραμμα πρέπει να ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει συγκεκριμένα, ξεκίνησε μάλλον συγκεκριμένα με το ΠΔΛΤΑΠΗ 1420 Πρόκειται για την ενσωμάτωση του υφισταμένου προγράμματος σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης. πλέμιση λοιπόν της απάτης και της παρατυπίας. Πρέπει να αυξήσουμε τις συνέργειες και την ευελιξία σε συνδυασμό με την απλούστευση των κανόνων. Υποβάλλω συναφώς τροπολογίες που θα υποβάλλουμε στην Επιτροπή Κόντ, που είναι η καθήλυνα αρμόδια. Θυμίζω επίση το ψήφισμά μα 3 Μαου 2018 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη ε, Ένωση και για του οικονομικού κανόνε, του δημοσιονομικού κανόνε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιολογούν το νέο πρόγραμμα. Πολλοί είναι γνωστοί, άλλοι αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το πρόγραμμα έχει ένα προπολισμό για την περίοδο 27 σε τρέχουσες τιμές και κάναμε κάποιους υπολογισμού για να δούμε σε τι μεταφράζονται λεφτά σε σταθερές τιμές 2018 σε υποχρεώσεις και πληρωμές. Για τα τρία επιμέρους ε, στοιχεία του προγράμματος κάναμε τους ίδιους υπολογισμού. Κάναμε λοιπόν όπως είπα υπολογισμού με βάση την ε, μέθοδο της μετατροπής κάποιων ε, θέσεων και γνωμών σε ποσά. Έκατα κλείδι. Διακείμεθα θετικό εναντί του νέου προγράμματο που προτείνει η Κομισιόν. Προσδοκούμε πραγματικά ότι στο πλαίσιο του επομένου ΠΔΠ το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί επαρκώ για να συμβάλλει με τρόπο ικανό στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Φερνάντες. Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον Τόμας που είναι σκιώδης, αλλά θα μιλήσω πορτογαλικά. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι ανάγκη δημοσιονομικός να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης. Το ποσό λοιπόν που βλέπουμε εδώ ουσιαστικά είναι ποσό που εξοικονομούμε γιατί καταπολεμούμε την απάτη. Γλιτώνουμε πολύ περισσότερα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο Σκιώδης δυστυχώς δεν είναι εδώ και ζητά συγγνώμη, κολλείεται. Ε, θέλω όμως να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του. Θα συνεργαστούμε περαιτέρω με τον εισηγητή. Η καταπολέμηση της απάτης, ξέρετε, απαιτεί αποτελεσματικότητα, απόδοση και διαφάνεια. Είναι όλα ουσιώδη. Και βεβαίως ο εισηγητής δεν πρέπει να ξεχάσει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλο της Όλαφ σε συνεργασία του βεβαίω με τα κράτη-μέλη. Θέλουμε επίση τα ποσά να εκφραστούν σε σταθερές τιμές και όχι σε τρέχουσες τιμές. Αυτό έχει ζητήσει και η Επιτροπή Προπολογισμών και το Κοινοβούλιο. Έχουμε υπεραμενθεί ανέκαθεν αυτή τη θέση. το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι ουσιαστικό. Χρειαζόμαστε επαρκή προπολογισμό εδώ για την απάτη για να προστατεύσουμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα τα συμφέροντα των πολιτών. Φυσικά, λέει πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Η κυρία Κορδιά Στάμπαλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι στην Επιτροπή αυτή δεν συζητάμε πολύ για το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της απάτης, όχι γιατί δεν είναι σημαντικό, αλλά γιατί τα χρήματα που πηγαίνουν εκεί είναι 160 εκατομμύρια για 7 χρόνια. Είναι ελάχιστο το ποσό αυτό. Όταν ε, μιλούσαμε για τις προτεραιότητες του πολιτούς δημοσιοκού πλαισίου, πάντα μιλάμε για τα μεγάλα ποσά. Οπότε τέτοια προγράμματα είναι προγράμματα το οποίο δεν συζητάμε. Θα έπρεπε όμως να εξετάσουμε την δυνατότητα αύξησης του ποσού του κονδυλίου για το πρόγραμμα αυτό. Έχει γίνει μελέτη 150 δισεκατομμύρια χάνουμε κάθε χρόνο μόνο από τις απάτες που γίνονται από το ΦΠΑ, έτσι, μόνο. Οπότε η γενική μας ε, συμφωνία δεν θα άλλαζε όσον αφορά τον προπολογισμό, δηλαδή αν διπλασιάζαμε το ποσό. Βάζαμε άλλα 160 εκατομμύρια. Γιατί τελικά αυτά που θα κερδίζαμε από τις απάτες που θα αποφεύγαμε θα οδηγούσαν σε απόσβεση του ποσού αυτού. Οπότε αυτή την παρατήρηση έχω να κάνω. Από εκεί και πέρα μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Ποιος άλλο θέλει το λόγο. Νομίζω ότι η απάτη διευκολύνεται λόγω του πληθωρισμού εθνικών νομοθεσιών, λόγω της πολυπλοκότητας των εθνικών νομοθεσιών, που δημιουργεί ακριβώ παραθυράκια για φορολογικά παιχνίδια. Ξέρουμε εταιρείε ε, γίγαντες της ψηφιακής τεχνολογίας όπως και οι δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρου στην Ευρώπη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είμαστε θύματα λοιπόν δικών μας αντιφάσεων. Έχουμε νομοθεσία για τον ιστορικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά με αρνητικό αποτέλεσμα. Και αυτό οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι το αντιλαμβάνονται. Πρόκειται για μια απαράδεκτη αντίφαση. Και αυτό πορεύει από την έλλειψη σύγκληση των εθνικών νομοθεσιών που προβαίνουν σε φορολογικό dumping, δημιουργώντας χάσματα, όχι παραθυράκια, χάσματα, τα οποία εκμεταλλεύονται τεράστιες εταιρείε. Και οι οποίε εν τέλει αξιοποιούν την νομοθεσία αυτή για να μην πληρώνουν το ευρωφόρο. Δίνω τον λόγο στον ισχυτή για να κλείσουμε. Όχι. Δεν έχετε κάποιο σχόλιο. Όχι. Πολύ ωραία. Κατάθεση τροπολογιών έως τις 12 το μεσημέρι 3 Οκτωβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 5 Νοεμβρίου. Λόγω στον κύριο Αλή και πάλι για την κοινή αγροτική πολιτική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. 1η Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την ρύθμιση της ε, στήριξης στρατηγικών σχεδίων που θα καταρτούν από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Εγγύσεων, το Γεωργικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτό για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην ε, γεωργία που είχαμε τα τελευταία χρόνια με τις τιμές ε, για παράδειγμα ε, όταν ανοίγονται ευρωπαϊκές αγορές στον κόσμο και για να τιμηθούν και οι νέες υποχρώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι στο κλιματικό και για να ανταποκριθούμε καλύτερα και στην γεωπολιτική κατάσταση. Απαιτούνται λοιπόν κάποιε αλλαγέ στην ΚΑΠ. Πρώτον πρέπει να εξυγχρονιστεί για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει αυτέ. Δεύτερον, η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να απλοποιηθεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτέ τι προκλήσει με το ελάχιστο δυνατόν κόστο. Και έπειτα πρέπει να υπάρχει και περισσότερη συνοχή με άλλε ευρωπαϊκέ. πολιτικές. Όσον αφορά λοιπόν αυτές τις διαπιστώσεις, χαιρόμαστε για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τι προκλήσει αυτέ με νομοθετικό πλαίσιο για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, επιπλέον από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να πιστήσω την προσοχή σας και σε άλλες τροπολογίες που θα μπορούσαμε να υποβάλουμε στην αρμόδια επί της Επιτροπή. Κάποιες από αυτές τονίζουν πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστασία των τροφίμων, αλλά και για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Τα πρότυπα πρέπει να διατηρηθούν. Έπειτα, πώς θα μειωθούν οι διαφορές μεταξύ χωρών μελών. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις περισσότερο απομακρυσμένες περιοχές, να στηρίξουμε τις οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις και τους νέους αγρότες. Προτείνονται διάφορες τροπολογίες λοιπόν όσον αφορά την χρηματοδότηση της ΚΑΠ ξεκινώντας από την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου του 2018 που συμπληρώθηκε από το ψήφισμα της 31ης Μαΐου 2018. Προτείνουμε 382,9 δισεκατομμύρια και 450 σε τρέχουσες τιμές για την επόμενη περίοδο. Και όσον αφορά τώρα τα δύο ταμεία, το Ταμείο Εγγύσεων και το Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε τις τροπολογίες 12 και 13 που αναφέρονται σε αυτό με τα ποσά. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της όσον αφορά ε, τα στρατηγικά σχέδια και τη στήριξή τους, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφάλεια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι το κείμενο αυτό έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιγητά. Ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρόταση αυτή, μια πρόταση την οποία μπορούμε να στηρίξουμε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή των συναδέρφων στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί εγκρίναμε μία θέση κατά της μείωσης η θέση μας δηλαδή ζητάει τη διατήρηση της χρηματοδότησης της κοινή γεωργικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, τουλάχιστον για τις πραγματικές τιμές 2014-2020 και να σεβαστούμε και τους γενικούς προσανατολισμούς. Η ΚΑΠ είναι ιστορική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πολιτική αυτή ε, πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει μια δυνατή πολιτική. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να στηρίξουμε το σύστημα των δύο πυλώνων, ε, εισόδημα πρώτος πυλώνας και ενισχύσεις δεύτερος πυλώνας. Όλα αυτά για το καλό των γεωργών αλλά και των καταναλωτών. Γιατί οι καταναλωτές χρειάζονται μια ασφαλή διατροφή και βιώσιμη. Σήμερα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια άλλη πρόκληση, την περιβαλλοντική μετά τη Συμφωνία των Παρισίων. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να επενδυθούν περισσότερα χρήματα για να ενισχυθεί αυτή η περιβαλλοντική διάσταση της γεωργίας μας. Αυτό λοιπόν που μας ε, απασχολεί και η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή σίγουρα θα ασχοληθεί περισσότερο, είναι τα νέα εθνικά στρατηγικά σχέδια πάνω στο οποία βασίζεται αυτή η πολιτική. Αυτά λοιπόν κάνουν διάκριση στις ε, πολιτικές των διαφόρων χωρών. Ενώ κατά το παρελθόν ακόμα και για τον πρώτο πυλώνα δεν συνέβαινε αυτό. Άρα δεν θα υπάρχει πια πραγματικά ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Θα έχουμε εθνικά στρατηγικά προγράμματα τα οποία θα εκπονεί η κάθε χώρα χωριστά. Ποιο είναι ο κίνδυνο, Ο κίνδυνο είναι ότι θα καταλήξουμε σε 27 διαφορετικέ ε, γεωργικέ πολιτικέ. Και έπειτα υπάρχουν και χώρε που έχουν ομοσπονδιακό χαρακτήρα με περιφέρειε, όπου και εκεί τελικά την αρμοδιότητα για τη γεωργία μπορεί να την αναλάβουν τα κρατήδια, οι περιφέρειες κλπ. Συνεπώ, από τη μια έχουμε το πλεονέκτημα της σύγκλησης ε, για μια γεωργική πολιτική πραγματικά ομοιόμορφη για όλες τις χώρες μέλη. Αλλά τώρα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινδυνεύουμε να βρεθούμε με 27 διαφορετικές γεωργικές πολιτικές. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προσέξουμε όλους ιδιαίτερος. Α υποθέσουμε ότι έχουμε δύο γεωργούς από την Μεσόγειο, από την ίδια περιοχή ελαιοπαραγωγού στην Ιταλία και στην Ισπανία. Θα μπορούσαμε να έχουμε δύο διαφορετικές πολιτικές στήριξης των εισοδημάτων στους, στις δύο χώρες. Γιατί στη μία οι ενισχύσεις θα είναι στεδεμένες, στις άλλες θα είναι κατά αποκοπή. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουν να βλάψουν την εσωτερική αγορά και κυρίως μια οι ενισχυσει θα ειναι στεδεμενες στι αλλες θα ειναι κατα αποκοπη ολα αυτα καταλαβαινετε οτι κινδυνευουν να βλαψουν την εσωτερικη αγορα και κυριως μια επιχειρηση η οποία ε, τελικά θα δουλεύει κάτω από συνθήκες αθέμη του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί με και εκεί συντάκτης γνωμοδότησης, φύγει αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι και η Επιτροπή Προπολογισμών πρέπει να καθορίσει προσανατολισμό. Και έπειτα υπάρχουν και τα θέματα της χρηματοδότησης που μας απασχολούν πιο άμεσα. Είναι αναγκαίο εδώ να επαναλάβουμε και να επιβεβαιώσουμε αυτό που πάντα κάναμε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εφόσον θα ετοιμάσουμε τη γνωμοδότησή μας γρήγορα, να πούμε ότι χρειάζεται κατάλληλη χρηματοδότηση για τη διατήρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής που όπως σας είπα πρέπει να είναι μια ισχυρή πολιτική και να επιτρέπει τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας σεβόμενοι το περιβάλλον, πράγμα το οποίο πετύχει μια παραπάνω προσπάθεια. Όταν λοιπόν ζητάμε παραπάνω προσπάθεια από τους γεωργούς μας, δεν μπορούμε συγχρόνως να τους μειώνουμε τις ε, ενισχύσεις. Συνεπώς πρέπει να προβλέψουμε το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης και εδώ νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα, η κυρία Γλουανέκ θα είχε κανονικά το λόγο, αλλά δεν είναι εδώ. Ωραία, κυρία Καρτσίνα Σαμπάλ. Ναι, οι συντονιστέ. Ε, αυτό, τι να κάνουμε. Σε μας πέφτει. Δύο σχόλια. Άκουσα τον κύριο Λαβία, που είναι ειδικό στα θέματα γεωργίας, αν και στον προπολογισμό δεν θα μπω στην ουσία, αλλά για την κοινή γεωργική πολιτική που είπε ότι είναι ιστορική σημασία. Πράγματι, Επιπλέον όμως είναι στην πραγματικότητα η μόνη ευρωπαϊκή πολιτική που είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκή. Και γι' αυτό πρέπει να δείξουμε. Είναι αλήθεια, έτσι. Ναι, σωστά. Και θα το πω και το απόγευμα, έτσι, όταν θα πάω για το Ταμείο Αλίας. Λοιπόν, έλεγα ότι πράγματι πρέπει να δείξουμε πόσο πολύ μας ενδιαφέρει η πολιτική αυτή και να μην δεχτούμε τις περικοπές που προτείνει η Κομισιόν. Αν υπάρχει μια σαφής γραμμή στο πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ακριβώς ότι δεν θέλουμε να αφαιρεθούν χρήματα από την κοινή γεωργική πολιτική. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Οπότε συμφωνούμε με τον εισηγητή. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η γεωργική πολιτική, αν δούμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι μία από τις πολιτικές που μπορεί να επηρεάσει, να βοηθήσει την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε την σημασία που έχει αυτή η πολιτική για την επίτευξη ακριβώς αυτών των στόχων. Θα συνεργαστεί η ομάδα μου με τον εισηγητή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλλος. Τότε θα ζητήσουμε από τον κύριο Σμικ να πάρει το λόγο. Γιατί εκείνος είχε αναλάβει τον ε, οριζόντιο κανονισμό ο κύριος Κουσμιούκ. Και υπάρχει σχέση ανάμεσα στην έκθεση του κύριου Αλή και την έκθεση του κύριου Κούσμιουκ. Γι' αυτό θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κούσμιουκ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, ήθελα οπωσδήποτε να το πω αυτό, διότι ε, ε, συμφωνώ με τα όσα άκουσα στο προηγούμενο σημείο και ακριβώς αυτά ήθελα να πω και εγώ για τη χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Λοιπόν, στην e, μείωση βλέπουμε στον πρώτο πυλώνα περίπου 32 δισεκατομμυρίων που ε, αντιστοιχεί σε 11% περίπου. Και 27 δις είναι η, μείωση ε, έτσι, με σταθερές τιμές, δηλαδή 28% για το δεύτερο πυλώνα. Αυτά τα πράγματα είναι τελείως απαράδεκτα. Σε μια κατάσταση όπως αυτή που ζούμε σήμερα, με επιπλέον απαιτήσει και επιβαρύνσεις για τους αγρότες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά και κλιματικά καθήκοντά τους. Άρα, ε, εδώ μιλώ για δύο ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαρτίου το ένα και το άλλο ήταν τέλη Μαΐου. γίνεται λόγος για τις πληρωμές από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για όλες τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές, για όλο το PDP. Είπαμε ότι θέλουμε η χρηματοδότηση να είναι 1,3% του ΕΠ. Αυτός να είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Πρέπει να είμαστε λογικοί και συνεπείς. Προτείνουμε ε, δαπάνες μιας συγκεκριμένη τάξεως ε, που θα πρέπει κάπως να καλύπτονται και στο ύψος των περιστάσεων και η κοινή γεωργική πολιτική με ένα ποσό τουλάχιστον συγκρίσιμο και αντίστοιχο του σημερινού. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα που είχα να πω για τη γεωργία. Έρχομαι τώρα στη δική μου γνωμοδότηση. Προτείνω και κάποιες άλλες λύσεις που μπορεί να είναι επίμαχες και να μην συμφωνούν οι συνάδελφοι, αλλά εγώ τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να καταργηθεί η διαφορά ανάμεσα στις άμεσες ενισχύσεις και τις υπόλοιπες, βασιζόμενη ε, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές της επόμενης περίοδου 2021-2027, ναι, ε, ε, θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την ένταξη τότε των 12 κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των λεγόμενων νέων χωρών. Τώρα θα πρέπει να θεωρούνται παλιέ και χώρε αυτέ, αυτές, γιατί οι επιχειρήσει λειτουργούν στην ίδια εσωτερική αγορά και υπακούν στου ίδιου κανόνε. Και οι γεωργοί σήμερα βρίσκονται σε δινή κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τι ε, ίδιε ηθίκε για όλους. Ε, κάνω και προτάσεις για το νέο γεωργικό αποθεματικό, που θα πρέπει να εγγραφεί χωριστά, κατά τη γνώμη μου, στον προϋπολογισμό. Ε, τα χρήματα του αποθεματικού αυτού δεν θα πρέπει να προέρχονται από τις άμεσες πληρωμές. Όπως ξέρετε, το αποθεματικό αυτό ε, έρχεται για να απαντήσει στους μηχανισμούς της αγοράς. Ενώ οι άμεσες ενισχύσεις έχουν άλλο σκοπό. Ε, θα παρακαλούσα να παραμείνουν τα πράγματα όπως έχουν σήμερα. Έχουμε ένα μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχία και για τους αγρότες μέχρι 2.000 ευρώ. Ε, αυτά θέλω να καταργηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρριγνύει τα ημάτια της για τη διαφάνεια και τη σαφήνεια και τη λειτουργία της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αλλά προτείνει γραφειοκρατικές ρυθμίσεις. Για τους μικρούς αγρότες όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν τα βγάζουν πέρα. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Είναι κάτι που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αυτόματη ανάκτηση των μη δαπανούμενων κονδυλίων. Ε, μιλώ για την, τις παρεμβάσεις στην Ήπεθρο. Διανύουμε τη δεύτερη χρονιά αυτού του μέτρου στο προϋπολογισμό και τώρα προτείνουν να καταργηθεί το νησιν 3 και να αντικατασταθεί από το νησιν 2. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό βελτιώνει πάρα πολύ τους, την κατάσταση των δικαιούχων. Το, το αντίθετο μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες προτάσεις που έχω στη γνωμοδότησή μου σε γενικές γραμμές. Είναι ίσως κάπως λιγότερο σημαντικές από τα όσα είπα στην αρχή. Μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Για να κλείσω θέλω να πω ότι στη συζήτηση για το προηγούμενο θέμα άκουσα όλες τις απόψεις των συναδέλφων και βλέπω ότι όλοι θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό ε, η ΚΑΠ να διατηρήσει τουλάχιστον τη σημερινή της χρηματοδότηση και να μην μειωθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα. Ο κύριος Φερνάντης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο σκιώδης ηγητής κολλείεται σήμερα και ε, ζητά συγγνώμη. Θα σας τα πω εγώ. Ευχαριστή επίσης τον εισηγητή. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι ένα success story. Έχουμε καλά τρόφιμα και ποιοτικά και ποσοτικά αρκετά προσβάσιμα. Αλλά τώρα ε, επιβαρύνουμε τους αγρότες με περιβαλλοντικά μέτρα. Ο σχέδιος ηγητής μας είναι πεπισμένος ότι αν δεν υπήρχε η κοινή γεωργική πολιτική θα ήταν τεράστιο το κόστος. Καμιά φορά τις πολιτικές ε, τις εκτιμάμε όταν τις χάνουμε, όπως και άλλα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν μια χρηματοδότηση σωστή έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υγιεινά και ε, ποιοτικά τρόφιμα που να σέβονται και περιβαλλοντικά πρότυπα και κανόνες. Κάτι που μας απασχολεί πολύ είναι η ανανέωση ηλικιακή δηλαδή της γεωργίας. Αν δούμε τη μέση ηλικία των γεωργών θα διαπιστώσουμε ότι είναι πολύ ψηλή. Αυτό δεν είναι άσχετο με την απόδοση της γεωργίας. Δεν συμφέρει να είσαι αγρότης. Τα άλλα επαγγέλματα αποφέρουν περισσότερο. Οπότε, κατά την άποψή μας είναι απαράδεκτες οι περικοπές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πολιτική συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιούσε για τους υπολογισμούς σταθερές τιμές. Αλλά στην κοινή γεωργική πολιτική, για να... Ε, κρύψει τις περικοπές έχει χρησιμοποιήσει τρέχουσες τιμές. Και σε τρέχουσες πυλές, στο, ε, ε, ε τιμές, στον πρώτο πυλώνα είναι 10% η ε, περικοπή, ενώ στο δεύτερο πάνω από 25%. Και αυτά θα πρέπει να διορθωθούν και να υπολογιστούν σε σταθερές τιμές. Επίσης, ο σκιώδης ηγητής μας θεωρεί ότι εκτός από τη χρηματοδότηση θα πρέπει να μειωθεί και η γραφειοκρατία. Και να μην πέσουμε στον πειρασμό επαναθνικοποίησης αυτής της επιτυχημένης, επαναλαμβάνω, πολιτικής. Για το νέο μοντέλο τώρα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, Είπαμε, πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία στα κράτη-μέλη, αλλά εκτός αυτού θεωρεί ο εισηγητής, ο σκιώδης εισηγητής μας, ότι το σύστημα ελέγχου που προτείνεται θα πρέπει να μπορεί να αναθεωρείται και ελπίζει να μην επιφέρει μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά ε, τους αγρότες. Πρέπει να απλουστεύσουμε την γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Υποθέτω ότι η κυρία Καρδία Σάβαλ θέλει το λόγο για να αντικαταστήσει τη συνάδελφό της, την κυρία Ρονέκ. Ναι, Πρόεδρε, αλλά ισχύουν τα προηγούμενα σχόλια και για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί το βασικό μήνυμα είναι ακριβώ ότι δεν θέλουμε κανένα είδου περικοπή στη γεωργική πολιτική. Κύριε Αλή μου, vous faire euh, Κύριε Κούσμιουκ, μάλλον. Να κάνω κι εγώ κάποια προσωπικά σχόλια για την ανάγκη διατήρησης των πιστώσεων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Όλοι μιλούν για ένα ευρωπαϊκό αγαθό, κοινό αγαθό ευρωπαϊκό. Ένα από τα αγαθά αυτά είναι η ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική, όπως είναι και η αλληλεγγύη με την πολιτική συνοχής. Βεβαίως χρειάζεται απλούστευση των διαδικασιών. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε στη χώρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά αν μιλήσετε με έναν αγρότη, που σε ρωτάει πώς λειτουργεί η κοινή γεωργική πολιτική. Ε, αυτό είναι επικίνδυνη αποστολή. Μια πολιτική που δεν μπορείς να την εξηγήσει δεν είναι πια πολιτική. Άρα ε, υπάρχει απέτηση βεβαίως διαφύλαξη, διατήρηση των πόρων στο ίδιο επίπεδο, αλλά και απλούστευση. Γιατί θα πρέπει οι αγρότες να έχουν και ένα εισόδημα. Και ένα προβλέψιμο εισόδημα. Αλλιώς, ποιος νέος θα θέλει να πάει να γίνει αγρότης. Και πού θα βρουν επενδύσει και χρηματοδότηση. Το εισόδημα του αγρότη όμως δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά και από την πολιτική ελευθέρων συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καμιά φορά διαπιστώνω ε, αντιφάσεις. Τι νόημα έχει να δίνουμε επιδοτήσεις στους βοοτρόφους εάν του οδηγούμε σε πτώχευση γιατί κάνουμε ε, εισαγωγέ βοήου κρέατο ε, από τις συμφωνίε που έχουμε με το Μερκοσούρ ή με το Μεξικό. Επίσης καμιά φορά σκέφτομαι ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και οι αλυσίδες διανομής λαμβάνουν υπόψη τις ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωση και τι σημαίνουν αυτές για το εισόδημα των αγροτών και συμπιέζουν προ τα κάτω τι τιμέ παραγωγού. Δηλαδή έχουμε ε, ένα είδος υπεξαίρεσης, εισφετερισμού των ε, πληρωμών αυτών από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Άλλο θέμα, η ποιότητα. Αυτό έχει να κάνει και με την ε, επισητιστική ε, ασφάλεια και κυριαρχία στην Ευρώπη. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα οι αγρότες μας να μπορούν να απαντούν και σε αιτήματα της κοινωνίας, σε σχέση με το κλίμα, σε σχέση με το περιβάλλον, την ευζοία των ζώων. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε την έρευνα. Τι νόημα έχει να καταργούμε κάποια φυτοφάρμακα εάν δεν υπάρχουν υποκατάστατα. Υπάρχουν κανόνες, αλλά θα πρέπει αυτοί να εφαρμόζονται παντού στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δημόσια λοιπόν κονδύλια που δίνονται στους αγρότες ε, ε, είναι το αντιστάθμισμα των ε, διάφορων, διάφορων υποχρεώσεων που επιβάλλουμε στους αγρότες για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ή στις προσδοκίες της κοινωνίας. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, στον παρόντα εισηγητή, γιατί άλλος αποχώρησε, για να κλείσει. Ευχαριστώ και εσά, Πρόεδρε και τους συναδέλφους, για την υποστήριξη. Χαίρομαι που ζητάτε περισσότερες πιστώσεις. Η Επιτροπή Άγκρη σίγουρα θα σας περιβάλλει με ενθουσιασμό όταν μάθει τα νέα. Διευκρινίζω ότι η έκθεση του κύριου Αλή, λέει ο Πρόεδρος, περιμένει τροπολογίες έως το μεσημέρι 3 Οκτωβρίου και κυρίω 5 ε, Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι κλπ. Γι' αυτά για τις δύο εκθέσεις. Ψηφίζουμε επίσης την Επιτροπή 5 Νοεμβρίου θυμίζω. Οπότε κλείσαμε με, με τις εκθέσεις επί διαφορών προγραμμάτων. Τελευταίο θέμα για σήμερα το πρωί είναι ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε. όσον αφορά το Ταμείο Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Λόγω των σοβαρών γεγονότων στην Πορτογαλία. Πρόεδρε, πρόκειται για αίτημα της Πορτογαλίας να κινητοποιηθεί το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για δύο εταιρείε οι οποίε ε, απέλησαν γύρω στους 1.200 εργαζομένους. Πρόκειται για υφαντουργικές βιομηχανίες, είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση, έξω και η υποψηφιότητα εντό εισαγωγικών συνολικό κόστος 7,7 εκατομμύρια ευρώ περίπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να καλύψει το 4,6 4,6 εκατομμύρια Πρόκειται για δομική διαρθρωτική εξέλιξη. Το σημαντικό προκειμένου είναι ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων που απολύονται για να μπορέσουν πιο εύκολα να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν επαγγελματική κατάρτιση και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να λάβουν αυτή την εκπαίδευση, αν γίνεται ακόμη και όσο έχουν τη δουλειά τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δρά λοιπόν και προληπτικά. Πρέπει όμως να παρέμβει και το Ταμείο Προσαρμογή στην ε, παγκοσμιοποίηση. Εκεί όπου, εάν και εφόσον τα άλλα ταμεία δεν έκαναν τη δουλειά τους. Χρειάζεται λοιπόν αντιστάθμιση των απολειών που υφίστανε αυτοί οι άνθρωποι έχοντα χάσει τη δουλειά του. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση είναι ένα συμπληρωματικό, αν θέλετε, ταμείο, συμπληρωματικό προ τα διαρθρωτικά και βεβαίω ε, προτιμούμε την πρόληψη, αν είναι δυνατόν, από τη θεραπεία, όπως λέμε και στην Πορτογαλία. Πρώτα να ευχαριστώ τον Χωσέ Μανουέλ για την έκθεσή του για τα δεινά τα οποία επισυμβαίνουν σε διάφορες περιοχές λόγω της μετακατάστασης μεγάλων παραγωγικών μονάδων. Όντως είναι καλό να εξασφαλίσει κανείς επανεκπαίδευση, αλλά κάθε φορά τρέχουμε να προλάβουμε όταν τα θύματα πλέον ανέρχονται σε εκατοντάδες λόγω απολύσεων. Γιατί κάθε μέρα κλείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσει άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Και έτσι, ναι, βέβαια. Σα συμφέρει να έχετε μεγάλη επιχείρηση και να την κλείσετε γιατί κάποιο θα παρέμβει και θα ενισχύσει. Αλλά για του άλλου ε, απολυμμένου, τίποτα. Εδώ είναι προφανέ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουν τα διαρθρωτικά ταμεία για να μην φτάνουμε σε απολύσεις και όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων να σβήσουμε τη φωτιά. Ξέρω όμως ότι σε πολλούς αρέσει το, το Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Το θέμα είναι να προσαρμοστεί ολόκληρη η Ευρώπη στην παγκοσμιοποίηση. Κατά προτιμήση πριν να φύγουν οι θέσεις εργασία να πάνε αλλού. Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία απειλεί θέσεις εργασίας, μέχρι και σε τράπεζες. Δείτε τα αποτελέσματα των τραπεζών, αστρονομικά κέρδη. Λοιπόν, θέλει τον λόγο, κύριε Φερνάντες, για να κλείσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, σιωπηρή συμφωνία. Ευχαριστώ τους αδέλφους που τη σιωπή τους συμφωνούν. Ε, χαίρομαι που η παρέμβαση μου, λέει ο πρόεδρος, ε, θεωρήθηκε σιωπή. Πολύ ωραία. Τροπολογίες. Προθεσμία κατάθεσης. 12 η ώρα 1η Οκτωβρίου. Ψηφορία στην Επιτροπή μας 8 ή 9 Οκτωβρίου και πάμε στην Ολομέλεια τη 2η του Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε τότε θα τα ξαναπούμε στις 2.30 διακόπτερη συνεδρίαση. Ε, χαίρομαι που τελειώσαμε νωρίς. Θα τα ξαναπούμε στις 2.30. Ευχαριστώ. <laughs> Et merde. Pardon.